Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να συνεχίσουμε. Η απογευματινή μας ημερήσια διάταξη είναι αρκετά ελαφριά, γιατί το πρωί προχωρήσαμε με ταχύς ρυθμούς και μεταξύ 12 και 2 συνεχίσαμε με τους συντονιστές τη συζήτηση για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012 και για τα θεσμικά όργανα, κοινοβούλιο και λοιπά τμήματα μετά την πολύ ενδιαφέρουσα και πλήρη ανταλλαγή απόψε που είχαμε το πρωί αλλά μιλήσαμε και για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνω τώρα να δώσουμε το λόγο στη Φραντσέσκα Μπαλτσάνη να μας ενημερώσει για τα συμπεράσματα που άντλησε από την πρωινή συνεδρίαση των συντονιστών. Και μετά, αν θέλουν οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο, θα τον λάβουν. Και αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, μπορούμε και να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Για το δημοσιονομικό κανονισμό τον έχουμε στην ημερήσια διάταξη, αλλά αν δεν έρθει εγκαίρος ο εισηγητής θα το αναβάλουμε για άλλη φορά. Έχουμε την ψηφοφορία άλλωστε για το δημοσιονομικό κανονισμό τη Δευτέρα. Κύριε Κοντμάνης, θέλετε το λόγο? Φραντσέσκα Βαλτζάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, έγινε μια μακροσκελέστατη συζήτηση στην ε, διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών και τα εκρεμή θέματα είναι ουσιαστικά τρία. Πρωτίστως, πριν από οτιδήποτε άλλο, πρέπει, διότι είναι πολύ σημαντική συνιστόσα του προπολογισμού μας, να κατανοήσουμε πώς θέλουμε να δούμε τις σχέσεις μεταξύ της χρηματοδότησης του ίτερ και της διαδικασίας του προπολογισμού μας. Η άποψή μας, την οποία σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζουν και οι συντονιστές από αυτή την πρώτη συνάντηση που είχαμε, είναι να είναι σαφής προτεραιότητα να έχουμε σε ε, συγκεκριμένο χρόνο τον προπολογισμό του 2012 αποφεύγοντας να έχουμε ε, παρεμβάσεις και καθυστερήσεις λόγω του τόσο ευαίσθητου ζητήματος του ίτερ. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι βαθύτατα πολιτικό και το να εντάξουμε την ε, χρηματοδότηση Twitter στον προϋπολογισμό μας ε, θα κάνουν ουσιαστικά διάφανες όλες τις προσπάθειες που κάνουμε για να έχουμε προτεραιότητες για τη στρατηγική για το 2020 και για την έρευνα. Διότι ε, αναφερόμαστε σε τελείως διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία. 540 εκατομμύρια για το ίτερ και έχουμε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ε, που χρησιμοποιούνται απλώς για τις υπόλοιπες ε, πηγές. Πρόκειται λοιπόν για ένα ενδιαφέρον ε, πρόγραμμα έρευνας και πολλές φορές είναι σημαντικό αυτό. Θα υπάρχουν επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό του 2020 αλλά εάν ενώσουμε τις δύο διαπραγματεύσεις και τις εξετάσουμε από κοινού, ελοχεύει ο κίνδυνος να μην έχουμε αυτό τον σταθερό και υπεύθυνο προπολογισμό που θέλουμε να έχουμε, διότι αναφερόμαστε σε χρηματοδότηση ε, μιας γραμμής προπολογισμού που με τα τόσα εκατομμύρια στα οποία θα διαθέσουμε εκεί φαίνεται ότι θα κάνει ε, αόρατα όλα τα υπόλοιπα που θέλουμε να έχουμε για το 2012. Επομένως, το πρώτο θέμα είναι να αποφασίσουμε να κάνουμε την πολιτική απόπειρα η χρηματοδότηση του Twitter να αποφασιστεί ξεχωριστά αφού θα έχει ολοκληρωθεί ο προπολογισμό, διότι είναι και κατεπήγον αυτό, είναι ένδειξη της σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο προπολογισμό το 2012. Υπάρχουν επίσης τομεί τομείς που είναι πολύ σημαντικοί, ε, ο Α και το τομέα 4 και οι τροπολογίε που παρουσίασαν οι επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πολιτικές ομάδες ε, θα έχουμε πολύ σημαντικές συνέπειες και θα αλλάξει ο προϋπολογισμός ε, ε, κατά 300 εκατομμύρια για το τομέα Α και για το τομέα 4 θα έχουμε αρνητικό ε, ψηφίο κατά 500 εκατομμύρια. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, ιδίως αυτούς τους δύο συγκεκριμένους τομείς. Ο τομέας 4 είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, διότι ήδη υπήρχε αρνητικό περιθώριο 153 εκατομμυρίων και λαμβάνοντα υπόψη και την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιλαμβάνει και τη διορθωτική επιστολή για τι χώρε τη Μεσογείου, ξεκινάμε ούτω ή άλλω με αρνητικό περιθώριο. Επομένω, οποιαδήποτε προσθήκη κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα, ε, απλώς επιδεινώνει την κατάσταση. Για τον τομέα λοιπόν 4 είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και αν θέλουμε μόνο να ε, σεβαστούμε τη θητεία, την εντολή που έχουμε ψηφίσει για τι τριμερεί συνομιλίε. Δηλαδή, να χρηματοδοτήσουμε τις χώρες της Μεσογείου και να κάνουμε ε, να λάβουμε υπόψη μας συγγνώμη και τη διορθωτική επιστολή και να έχουμε χρηματοδότηση για την Παλαιστίνη είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην μας οδηγήσει σε ένα σημαντικό αρνητικό περιθώριο. Υπάρχει και το θέμα των πληρωμών το οποίο είναι στρατηγική σημασίας αλλά και ουσιαστικό διότι Πρόκειται για το κινητήριο μοχλό ε, του προπολογισμού. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις υποχρεώσεων και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι πληρωμέ που μας δείχνουν πώς σεβόμαστε αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει χρονικά. Για τις τριμερεί ομιλίες έχουμε ζητήσει να λάβουμε υπόψη ε, ότι θα πρέπει να λάβουμε το τομέα αυτό ω ε, ένα ελάχιστο ποσό. το προσχέδιο του προπολογισμού και από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφοροι τομείς που είναι σημαντικοί. Υπάρχει η, ο τομέα είναι και για τι πληρωμές ε, ούτω ή άλλω θα είναι πολύ ευαίσθητα τα πράγματα στη διαπραγμάτευση. Τα όσα έχουμε ψηφίσει στην εντολή που δώσαμε για τη διαπραγμάτευση αποτελούν καλό σημείο εκκίνηση. Αυτά βέβαια είναι όλα υποθετικά σενάρια εργασίας. Οι τροπολογίες που παρουσιάστηκαν και από τα μέλη της Επιτροπής και από τις Επιτροπές και από τις πολιτικές ομάδες αποτελούν σημαντική πρώτη ύλη ώστε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε από εκεί και πέρα σε ισορροπημένες λύσεις ξεκινώντας από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα εγώ είμαι πολύ ανοιχτή και πραγματικά ελπίζω πολύ στις προτάσεις των πολιτικών ομάδων και των μελών της Επιτροπής μας, διότι η πρόκληση είναι να προσπαθήσουμε να εξέφουμε μια ισορροπία μεταξύ ενός προπολογισμού, ο οποίο έχει πολύ στενά περιθώρια, μιας εντολής που έχουμε ήδη ψηφίσει στην Ολομέλεια που μας δίνει κάποιε κατευθυντήρε γραμμές και της ανάγκη να δώσουμε ε, ένα, μια χρηματοδότηση στις προτεραιότητες που έχουμε καθορίσει. Και έχουμε πει επαναλημμένως ότι δεν είναι ανούσιες αυτές οι προτεραιότητες, αλλά είναι προτεραιότητες στρατηγικής του Ευρώπης του 2020 και αυτές πρέπει να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε. Ευχαριστούμε την συγχύτρια Τζοβάνι Λαβία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι από τα όσα μας είπε η συγγήτρια, την οποία και ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά που έκανε και κάνει ακόμα, διαφαίνεται σαφώς ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να τα δούμε ξεχωριστά. Η συγγήτρια αναφέρθηκε ε, προφανώς στη χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ συμφωνώ μαζί της, δεν μπορούμε να το δούμε αυτό από κοινού με το υπόλοιπο τμήμα του προπολογισμού. Είναι σαφές ότι ο τρόπος που ε, αντιλαμβάνεται το Συμβούλιο των Προπολογισμού και οι προτάσεις περικοπών ε, που σχετίζονται με το ε, κλείσιμο της ε, γεωργικής χρηματοδότησης ε, μας οδηγούν σε κάποια μετατόπιση των αποφάσεών μας γνωρίζουμε μεν πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό, αλλά η λύση για τη χρηματοδότηση του Ίτερ θα πρέπει να βρεθεί σε άλλη συζήτηση. Έχω την εντύπωση όμως ότι στο σημείο 1α θα πρέπει να εξετάσουμε ένα επιπλέον σημείο, μια προτεραιότητα την οποία ε, θελήσαμε εμείς ε, και μάλιστα με ιδιαίτερο σθένος στο Κοινοβούλιο και σχετίζεται με την ε, επανέναρξη μιας ε, ευρωπαϊκής οικονομίας η οποία βιώνει η κρίση αυτή τη στιγμή και τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε εκ νέου κάποια πράγματα. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε περικοπές στα πλαίσια του 7 προγράμματος πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε και μάλιστα σε γραμμές οι οποίες ε, σαφώς μπορούν να εφαρμοστούν. Τίθεται λοιπόν το εξής πρόβλημα όπως έλεγε και η συγγήτρια. Τι περιθώριο ελιγμών έχουμε στο συγκεκριμένο τομέα του προϋπολογισμού και ως προς αυτό θα πρέπει να γίνουν συνειδητές επιλογές. Συνειδητές επιλογές σημαίνει ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες στις οποίες θέλει να επενδύσει το Κοινοβούλιο, αλλά αφετέρου να είμαστε πάντα ρεαλιστικοί στην προσέγγιση που έχουμε προς τον προϋπολογισμό. Ρεαλιστική σε περίοδο κρίσης σημαίνει να μείνουμε εντός ενός πλαισίου χρηματοδότησης, το οποίο θα είναι συμβατό με το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιπλέον αντιπαραθέσεις για το σημείο αυτό, διότι αυτό το οποίο προέκυψε από τις τροπολογίες που παρουσίασαν οι επιτροπές και οι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, ελοχεύει ο κίνδυνος να ξεπεράσουμε κατά πολύ το ανώτατο όριο δαπανών της κατηγορίας αυτής και νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα τέτοιο στόχο. Επιπλέον, το άλλο πρόβλημα συνδέεται σίγουρα με την κατηγορία 4. Η κατηγορία 4 είναι μια κατηγορία στην οποία ήδη και στο παρελθόν είχαμε υπερβεί το ανώτατο όριο δαπανών, ε, χρησιμοποιήσαμε τη δυνατότητα της ευελιξίας και πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ευρωπής ε, είχε λάβει υπόψη της ε, σωστά ορθώς τις δαπάνες. Στον, ε, στην κατηγορία 4 λοιπόν οι προτάσεις που κάνουν οι αρμόδιες επιτροπές μας φαίνουν πολύ πέρα από το ανώτατο όριο δαπανών και νομίζω ότι με τους ε, των επιτροπών ΔΕΒΕ και ΑΦΕΤ θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο εις βάθος το ζήτημα για να επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες. Η προτεραιότητα της Μεσογείου είναι η μία και ήδη πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες προφανώς, τις οποίες έχουν εντοπίσει οι αρμόδιες επιτροπές και πρέπει να τις εντοπίσουν οι αρμόδιες επιτροπές. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Το θέμα των πληρωμών είναι σημαντικό, αλλά είναι και δύσκολο και για το Συμβούλιο και για τα κράτη-μέλη σε περίοδο κρίσης και είναι σίγουρα το σημείο το οποίο θα παρατηρήσει το Συμβούλιο, θα προσέξει το Συμβούλιο περισσότερο στη συνδιαλλαγή. Υπάρχει επίσης ε, ο τομέας 1β. Εκεί προβλέπεται να υπάρχει μια χρηματοδότηση και μια πρικοδότηση η οποία θα είναι επαρκής για την, ε, ε, με βάση τον προϋπολογισμό. Η Αποκατάσταση λοιπόν κάποιων γραμμών προπολογισμού όπω ζήτησαν οι αρμόδιε επιτροπέ είναι απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν επίση κάποιε άλλε προτεραιότητε τι οποίε θα πρέπει να καθορίσουμε και θα ήθελα να επιγραμμίσω ένα ζήτημα για το τομέα 2, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για αρκετέ πολιτικέ ομάδε, καθότι κατέθεσαν τροπολογία ε, πολλέ πολιτικέ ομάδε. Δεν υπάρχει νομική βάση για το σημείο αυτό και νομίζω ότι στη συνδιαλλαγή θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει μία προσαρμογή που θα δίνει και μία ε, θετική πτυχή της Ευρώπης προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μία τόσο δύσκολη περίοδο κρίσης, στην οποία αυξάνονται οι άνθρωποι που έχουν ανάγκες, να ε, γίνουν περικοπές ε, στο Ταμείο για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο. Το ο κύριος Γκοτμάνης. Θα ήθελα να επισημάνω τρία σημεία. Το πρώτο αφορά τη στρατηγική του Συμβουλίου ε, για το πρόγραμμα των εξαμήνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει 13% ε, για τις πληρωμές και 17% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Σημαντικά. Ενώ το Συμβούλιο είπε 7,5% για τα για τι πληρωμέ και 6,7 για, για την ανάλυση υποχρεώσεων. Το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα Πελέσιο έχει υποδιπλασιαστεί από το Συμβούλιο προ τον προπολογισμό του. Και μερικές φορές, όπως μας είπε ο κύριος Λεβαντόφσκι, υπάρχει πρόβλημα με ορισμένα προγράμματα γιατί δεν προχωρούν. Οπότε, γιατί να έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό αύξησης. Αλλά θέλουμε μία ξεκάθαρη απάντηση. Ισχύει αυτό ή όχι, γιατί η Γενική Διεύθυνση Έρευνα λέει ότι φέτο δεν πρόκειται να απορροφηθούν όλοι οι πόροι, όλα τα κονδύλια. Άρα υπάρχει ε, αντίφαση. Από την μια προτείνει μεγάλη αύξηση, από την άλλη είναι ανικανότητα φαίνεται απορρόφηση. Δεύτερον, ε, στις πληρωμές έχουμε 3% αύξηση την Γεωργία. Τώρα φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας ε, της σταδιακής ένταξης, όπου οι χώρες θα πληρώνουν περισσότερο. Και παρόλα αυτά, το Συμβούλιο τα έκοψε στη μέση, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί και πού βρίσκεται αυτό το αποθεματικό, δεν είναι σαφές. Φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας Facing ε, in, σταδιακής ένταξης, σταδιακής εισαγωγής. Πού σκοπεύει το Συμβούλιο να αφιερώσει τα κονδύλια αυτά. Και η τρίτη ερώτηση που είναι πιο μακροσκελής. Έλαβα τα τελευταία στοιχεία στις 13 Σεπτεμβρίου για την απορρόφηση των κονδυλίων συνοχής στις 27 χώρες μέλη. Είναι πρόσφατα στοιχεία, μια εβδομάδα πριν τα έλαβα. Αν ρίξετε μια ματιά στην πρόταση για τα κονδύλια της συνοχής, τι διαπιστώνετε. Διαπιστώνετε δύο τινά. Πρώτον, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο το Συμβουλίο, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να μειώσει τις πληρωμές και μάλιστα δραστικά και φέτος πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές. Μείον 30% πληρωμές φέτος σε σχέση με πέρυσι για τη διάσταση περιφερειακής ανάπτυξης στο Ταμείο Συνοχής. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι χώρες που είναι επιλέξιμες και υπεύθυνε για να τα απορροφήσουν αυτά είναι συνήθως οι παλιές χώρες, γιατί οι νέε χώρε δεν εμπίπτουν σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι παλιέ χώρε δεν θα μπορέσουν φέτο να απορροφήσουν τα απαραίτητα κονδύλια. Και επιπλέον το Συμβούλιο επέτεινε αυτέ τι περικοπέ πρότεινε ακόμη πιο δραστικές περικοπές. Ένα δις περίπου περικοπέ. Πολύ σοβαρό αυτό. Και αν είχαμε στο σχέδιο πληρωμές συν 6% η ε, μείωση είναι 3%. Είναι τόσο κακή η εφαρμογή. Αν μια ματιά στα στοιχεία εφαρμογής της 14 η Ιουνίου, πριν από δύο μήνες δηλαδή, για την εφαρμογή ε, του προγράμματος, περίπου έχει περάσει ένα εξάμεινο και βλέπουμε ότι για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή μάλλον συγγνώμη διορθώνε μιλητής, για το Κοινωνικό Ταμείο είναι αλήθεια ότι η διάσταση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας έχει υλοποιηθεί μόνο κατά 14% αλλά η σύγκληση κατά 44%. Δηλαδή για το κοινωνικό ταμείο τα στοιχεία μας δείχνουν μέσα σε ένα εξάμεινο οι χώρες που ε, απορροφούν ταμεία από το Κοινωνικό Ταμείο για την περιφερειακή ανάπτυξη, περιφερειακή συνεργασία δεν ε, έχουν καλούς ρυθμούς και η Επιτροπή είναι απεσιόδοξη. Πέρυσι είχαμε 13% ε, απορρόφηση, την ίδια ημερομηνία, 14 Ιουνίου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εκεί η σύγκληση, για τη σύγκληση, Έχουμε 37% εκτέλεση. Μικρές οι διαφορές λοιπόν. Οπότε το Συμβούλιο μειώσει επιπλέον, κόψει επιπλέον ένα δισεκατομμύριο από την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, δεν ξέρω πού στηριχθήκατε για μια τέτοια πρόταση. Τι βάση δεδομένων χρησιμοποίησατε. Και τέλος, αν ρίξετε μια ματιά στα κονδύλια αυτά, στα νούμερα αυτά, ξέρω ότι θα υποβληθούν και άλλες προτάσεις δεν θα επεκταθώ. Μία και μόνο ερώτηση έχω. Αν αναλύσετε τι διαφορέ μεταξύ των διαφόρων χωρών σήμερα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων, διαπιστώνουμε ότι οι διαφορέ εξακολουθούν να είναι σημαντικέ. Στο Περιφερειακό Ταμείο 3,4 η καλύτεροι είναι οι καλύτεροι μαθητέ είναι πολύ καλύτεροι από του χειρότερου, κατά 3,4. 41% βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο. Και αν δούμε τι διαφορέ μεταξύ παλιών και νέων χωρών, διαπιστώνουμε τις ίδιες διαφορές. Μερικές νέες χώρες είναι δυόμιση φορές χειρότερες από τις καλύτερες χώρες και οι παλιές 15 χώρες έχουν διαφορά τριπλάσια. Υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης δηλαδή. Πάντως πολύ φοβούμαι ότι αν γίνει μια οριζόντια περικοπή και αν έχουμε ένα κριτήριο για όλους, γιατί ακόμη και μεταξύ παλιών και νέων χωρών έχουμε μερικές που είναι πολύ καλές και στις νέες και στις παλιές. Και δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε τις χώρες αυτές λέγοντας Γενικώ υπήρχε μικρή απορρόφηση, κόψτε ένα δισεκατομμύριο γιατί δεν θα υπάρξει δυνατότητα απορρόφησης. Είμαι μέλος τη Επιτροπής ε, περιφερειακή Ανάπτυξης και γνωρίζω του υπαλλήλου τη ε, Γενικής διεύθυνση ε, Ρέγγι και μου είπαν ότι πολύ καλά δουλεύουμε, είναι, καλά τρέχουν όλα τα προγράμματα. Βέβαια έχουμε κρίση, έχουμε συγχρηματοδότηση και η ανάπτυξη πέθριου είναι λίγο προβληματική. Αλλά θα ήθελα να εκφράσω τις σοβαρές μου επιφυλάξεις και να θέσω μια ερώτηση. Είναι σωστό το μήνυμα αυτό δεδομένων των χαλεπών καιρών. Μια οριζόντια ανάπτυξη, ε, περικοπή χωρίς κριτήριο, οπότε ουσιαστικά θα πλήττουμε ε, τους καλούς μαθητές, μια και δεν θα λαμβάνουμε υπόψη και δεν θα τους επιβραβεύουμε. Ευχαριστώ, συνάδελφε, και σας ευχαριστώ για τον πολύ σχολαστικό έλεγχο που κάνετε και για, τις, τα ποσοστά απορρόφησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε κυρία Μπαλτσάνη για την έντιμη και καλή εργασία που έκανε, της συνθέσεως δηλαδή. Και εμείς συμφωνήσαμε ότι το ίτερ πρέπει να μείνει εκτός των συζητήσεων. Είναι σημαντικό το θέμα και θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό του 2012. Η πολιτική μου ομάδα το στηρίζει το έργο αυτό, δεν είμαστε αντίθετοι. Θέλουμε να εκτελεστεί, αλλά όχι σε βάρος του 7ου προγράμματος πλαισίου. Άρα τα χρήματα να μην δαπανηθούν από την έρευνα. Θα πρέπει να βρεθεί λύση εκτός των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν χρήματα στον φετινό γεωργικό προϋπολογισμό που θα μπορέσουν να μεταφερθούν. Ελπίζουμε. Σε ό,τι αφορά τους άλλους τομείς του 1α, η πολιτική ομάδα έχει υποβάλει ορισμένες τροπολογίες που επανέρχονται στην πηγή, αλλά και παραπέρα, σχετικά με τους νέους οργανισμούς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά νομίζουμε ακόμη ότι υπάρχει ανάγκη να επανεξεταστούν ορισμένα κονδύλια της έρευνας που δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά, αλλά υπάρχουν και άλλα κονδύλια τα οποία έχουν πολύ καλή εκτέλεση και επίσης και η ενέργεια που για μας είναι μεγάλη προτεραιότητα. Και αν σημαίνει ότι πρέπει να υπερβούμε την οροφή, ας την υπερβούμε, τουλάχιστον ως διαπραγματευτική θέση. Το ίδιο για την κατηγορία 4, όπου έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες και ιδίω να υπάρξει μια δίκαιη λύση για το Παλαιστινιακό. Όπως είδαμε και στην πρόταση της Κομισιόν, θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό ευελιξίας, το εργαλείο ευελιξίας και αυτό θα πρέπει ίσως να κάνουμε. Για τον γεωργικό προϋπολογισμό, για το Συμβούλιο δηλαδή, του προϋπολογισμού Γεωργίας έχουν μάλλον επιλέξει ένα περίεργο τρόπο δράσεως διερωτώ και θα ήθελα να μάθω γιατί διότι ίσως το Συμβούλιο δεν σκέπτεται παρά μόνο ένα ποσό δηλαδή το ποσό των πληρωμών και δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς θα μπορέσουν να κάνουν πραγματικές περικοπές που είναι δύσκολο βέβαια Εάν γίνουν όμω περικοπές στα αγροτικά θα πρέπει να γίνουν με ευφιέστερο τρόπο. Και αυτό είναι δύσκολο. Με την αγροτική πολιτική όπως είναι τώρα, με τι μοναδικέ πληρωμές. Είναι δύσκολο να καταγραφούν ξεκάθαρα οι ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν και, υπάρχει το Ταμείο για την διανομή τροφίμων στους ε, φτωχούς ανθρώπους που πλέον δεν έχει νομική βάση. Ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια υποκατάσταση της βάσης αυτής. Ελπίζω στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να υπάρξει. Δεν έχουμε βέβαια τα αποθέματα βόλου κρέατος και άλλων που είχαμε παλαιότερα. Βρισκόμαστε σε διαφορετική κατάσταση τώρα και αυτό σημαίνει βέβαια ότι υπάρχουν και λιγότερα χρήματα διαθέσιμα στο κονδύλιο. Ο κ. Κοντμάνης μίλησε για την εφαρμογή και απορρόφηση στο 1β. Και εδώ βλέπουμε να κάνει περικοπές στο Συμβούλιο διότι επιθυμεί να καταλήξει σε ορισμένο ποσό των πληρωμών. Η κυρία Μπανζάνη θύμισε το έγγραφο που συζητήσαμε και εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο πριν από το καλοκαίρι, να μην δεχθούμε δηλαδή τέτοια περικοπή. Ωστόσο η πολιτική μου ομάδα έχει εκφράσει κάπως διαφορετική θέση. Εμείς θέλουμε το πλεόνασμα το περσινό να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί εις ώστε η περικοπή να είναι μικρότερη. Και αν το Συμβούλιο δέχεται μικρότερη περικοπή, γιατί όχι. Δεν μπορούμε τώρα να πάρουμε το πλεόνασμα του περσινού χρόνου. Αλλά μήπω μπορούμε να πάρουμε από το πλεόνασμα του επόμενου χρόνου. Διότι πάντα υπάρχει πλεόνασμα. Δεν δαπανώνται όλα τα κονδύλια και κυρίω κυρίως αυτά που μαρκάρονται για τα διαθωτικά ταμπία. Αυτό θέλω να εξεταστεί. Και όχι επειδή θέλουμε κάποια χώρα να δούμε να χάνει και να μην λαμβάνει τα χρήματα που τις αξίζουν, που χρειάζεται, αλλά όταν ολοκληρώνεται ένα έργο πρέπει να γίνει η πληρωμή και αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο κονδύλιο τότε το Συμβούλιο πρέπει να προβλέψει νέα χρήματα και αυτό είναι που δείχνει πόσο ανόητη είναι η θέση του Συμβουλίου που εμένει σε ένα ποσό αλλά αυτό είναι που θέλουν και αυτό ίσως μπορεί να μας επηρεάσει Τέλο πάντων α έχουν το ποσό που θέλουν αλλά όχι σε βάρος της έρευνα. εάν υπάρξουν, αν είναι να υπάρξουν περικοπές α υπάρξουν περικοπέ, εκεί όπου έχουν δικαίωμα να εισπράξουν τα χρήματα οι χώρες μέλη αλλά ας αποκαλύψουμε τον ανόητο τρόπο με τον οποίο εκτελείται η πολιτική αυτή θα πρέπει να μείνουμε αυστηρά στις προτεραιότητές μας για τον στόχο του 2020. Ευχαριστούμε. Αν σαφέστατα. Ο κύριος Μούλντερ. Ευχαριστώ. Μιλάνε όλοι φιλελεύθεροι εδώ, αλλά τέλος πάντων. Α, ήρθατε κι εσείς. Εντάξει. Έχω να προσθέσω κι εγώ κάποια πράγματα σε αυτά που είπαν μόλις οι συνάδελφοι. Καταρχάς, η αύξηση στις ε, πληρωμές. Στη χώρα από την οποία κατάγομαι, ελέγχθη ότι υπάρχει ανευθυνότητα από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλουν αύξηση στον προπολογισμό άνω του 4%. Όλε οι χώρε, συμπεριλαμβανομένε και των κάτω χωρών, πρέπει να κάνουν περικοπέ. Και μπορεί κάποιος να πει εκατοντάδες φορές ότι μπορεί να είναι συνέπεια προηγούμενων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι χώρες μέλη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρώνει ε, τις υποχρεώσεις της. Ε, αυτή την άποψη έχω εγώ για τις πληρωμές. Τώρα, ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων, ένα από τα βασικά σημεία νομίζω που είναι σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα ε, υπόλοιπο προς εκαθάριση άνω των 200 εκατομμυρίων και πολλοί λένε ότι αγγίζει και τα 250 εκατομμύρια ευρώ δισεκατομμύρια συγγνώμη, ευρώ. Ε, πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε ότι μπορούμε να έχουμε αυξημένες αναλήψεις υποχρεώσεων και απ' την άλλη έχετε και ένα υπόλοιπο προσεκαθάριση που είναι τετραπλάσιο του προπολογισμού του Ταμείου Συνεχής. Εξού λοιπόν και η πρόταση της Αν Γιάνσεν και η δική μου ζητάμε το 10% των υποχρεώσεων να μπουν στο αποθεματικό, μόνο στο αποθεματικό, που σημαίνει ότι τηρούμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά προς το παρόν θα μπουν στο αποθεματικό και θα ήθελα να υπάρχει και μια σαφής ανάλυση για το πώς αυτό το υπόλοιπο προσεκαθάριση είναι πάντα τόσο υψηλό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει τα στοιχεία, να μας πει ε, πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Ε, τι γίνεται με τους κανόνες νησιν 1, νησιν 2 και τις προηγούμενες αναλήψεις υποχρεώσεων. Πού προκύπτει το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ε, και καλή ε, έξωθεν μαρτυρία προς το ευρύ κοινό ότι ε, τηρούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει και στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς μπορούμε είτε να τα βγάλουμε από το θεματικό ή να ζητήσουμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό αν θεωρηθεί απαραότητα εν ώψη των νέων μέτρων αλλά θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις αναλήψεις υποχρεώσεων διότι κατά την άποψή μου είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στο ευρύ κοινό ε, πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτές τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις και την άλλη ένα τεράστιο ποσό το οποίο δεν μπορούμε να δαπανίσουμε. Ευχαριστούμε, ο κύριος Βόγκαν. Ευχαριστώ. Καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολες θα είναι οι διαπραγματεύσεις. Παρόλο που το Συμβούλιο συμφώνησε για αύξηση στις πληρωμές 2,2%, πολλές χώρες είπαν ότι αυτό είναι υπερβολικό. Και Ορισμένες χώρες θα δώσουν πραγματικά μάχη ε, και το χρησιμοποιούν αυτό κυρίως για ισοκομματικούς λόγους, ε, αλλά θα είναι δύσκολες οι πειραγματεύσεις σίγουρα. Το Συμβούλιο εξέτασε σοβαρά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτές που αποκαλούμε off-book και ορισμένες χώρες είπαν ότι η αύξηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι 5%, είναι ουσιαστικά 10% εξαιτίας της πρώτης softbook. Και αυτό θα είναι πρόβλημα στη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο. Πάντως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ιδιαίτερα να ε, φιλοδοξία να δείξουμε στις δημοσιονομικές γραμμές που προωθούν ε, απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτική συνοχή, ε, καινοτομία, τεχνολογική ανάπτυξη, υποδομέ. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι τομεί θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια να βρούμε τρόπου για να προωθήσουμε και δημοσιονομικέ γραμμέ στο κεφάλαιο 1α, γιατί αυτέ ε, έχουν δυναμικό δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα ήθελα όμω να προστατεύσουμε και το 1β και εδώ διαφέρω από του άλλου φιλελεύθερου συναδέλφου μιλήσαμε για τα διαρθρωτικά ταμεία και τη συνοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως έχουμε προβλήματα απορρόφησης, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουμε αυξημένο ρυθμό απορρόφησης. Στην Ουαλία, για παράδειγμα, τη γενέτειρά μου, περίπου 80% των διαρθρωτικών κονδυλίων έχουν ήδη απορροφηθεί και μερικά κονδύλια έχουν εξαντληθεί. Θα ήταν λάθος να περιορίσουμε τις αναλήψεις υποχρεώσεων στα διορθωτικά ταμεία και στη συνοχή. Αν θέλουμε οικονομίες να τις κάνουμε αλλού και όχι στις δημοσιονομικές γραμμές που προωθούν οικονομική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Όπως είπε η Αν θέλουμε να προστατεύσουμε το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο, να βγάλουμε το ίτερ. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε και το κενό ώστε να προασπίσουμε και την χρηματοδότηση Twitter στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την ελαστικότητα. Πέρυσι ζητήσαμε ελαστικότητα και το χρησιμοποίησαμε ως επιχείρημα με το Συμβούλιο. Θέλουμε ελαστικότητα στον προπολογισμό. Είπαμε να συνεχίσουμε το αποθεματικό, αλλά πέρυσι δεν προχωρήσαμε πολύ σε αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα ελαστικό, ε, ευελιξίας. Το ίδιο το μέσο ευελιξίας, για παράδειγμα. Γιατί να μην ε, διεκδικήσουμε ένα πιο ευμεγεθές τέτοιο μέσο ευελιξίας. Αυτό θα μας εξασφαλίσει ελαστικότητα στον προπολογισμό. Ξέρω ότι διαφωνούμε το Συμβούλιο για άλλα στοιχεία ευελιξίας, αλλά ίσως για το μέσο ευελιξίας καθ' αυτό δεν θα έχει μεγάλο πρόβλημα το Συμβούλιο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα αυτή την πορεία να ακολουθήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Βόν. Ο Γκέραν Φέρμ. Ε, <clears throat> ε, Ευχαριστώ. Και και την εισηγήτρια που μας έχει υποβάλει και ορισμένες επιλογές και όχι μόνο μία πορεία προς τα εμπρός. Πάντως πρέπει να συζητήσουμε και στην Επιτροπή μας ποια επιλογή θα επιλέξουμε. Είναι παρόμοια πάντω η ανάλυση μα, έστω και αν έχουμε αρισμένε διαφορέ ανάμεσα στι πολιτικέ ομάδε, αλλά δεν απέχουμε και πολύ. Όλοι προτιμούμε μια επιλεκτική προσέγγιση. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα αυξήσουμε όλα. Ουδή ζητεί ευρύτερη αναθεώρηση του πλαισίου. Θέλουμε να εμείνουμε στο εργαλείο ευκαμψίας. Οι ίδιες προτεραιότητες για το 1α και το 1.4. Οι διαφορές είναι πρώτο το επίπεδο φιλοδοξίας. Θα ακολουθήσουμε το πιο σόφρον πρότυπο που προτείνει η εισηγήτρια ή τα πιο φιλόδοξα για, την, ε, για τον τίτλο 4 και ίσως υπάρξουν ορισμένες διαφορές προτεραιοτήτων σε ορισμένα κονδύλια, αν και για παράδειγμα η διαβίου κατάρτιση η η Παλαιστίνη στο 4 στην ουσία είναι στόχοι που μοιράζονται όλες οι ομάδες. Δεν απέχουμε πολύ λοιπόν. Η διαφορά που βρίσκεται. Η δική μου πρόταση θα είναι να επιλέξουμε τις πιο φιλόδοξες προσεγγίσεις και στην κατηγορία 1α και στην κατηγορία 4. Πρώτα-πρώτα το ζήτημα είναι πολιτικό και είναι απαραίτητο για μας να επιτύχουμε πρόσθετες πληρωμές, κυρίως για την απασχόληση, για πολιτικές απασχόληση. Αυτό είναι σημαντικό για την οικονομία της Ευρώπης και πρέπει να δείξουμε και τι κάνουμε με τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, που είναι σημαντικό για την Ευρώπη και είναι σημαντικό να, είμαστε, να φανούμε φιλόδοξοι, γιατί πρόκειται για επενδύσεις στο μέλλον της οικονομίας μας και στο μέλλον της απασχόλησης. Αυτό είναι ο βασικός λόγος. Το ίδιο ισχύει και για την σημασία της πολιτικής γειτονίας και για την Παλαιστίνη στην κατηγορία 4. Βέβαια, είναι και κίνηση τακτικής, διότι το πρόβλημα είναι εάν αρχίσουμε από την λιγότερο φιλόδοξη προσέγγιση, ο κίνητος είναι να φτάσουμε στο μηδέν. Αν ξεκινήσουμε πιο φιλόδοξα, έχουμε την πιθανότητα να καταλήξουμε σε κάτι, έστω και αν είναι λιγότερο, φιλόδοξο. Για αυτό το λόγο εμείς επιλέγουμε την πλέον φιλόδοξη προσέγγιση και για το 1α και για το 4. Δεν θα σχολιάσω περισσότερο για το ίτερ. Έχουμε συμφωνήσει στη στρατηγική. Μία ερώτηση προς την Κομισιόν και ίσως και προς την εισηγήτρια. Γνωρίζουμε ότι το θέμα των πληρωμών είναι κρίσιμο και πολύ ευαίσθητο για τις χώρες μέλη. Η Κομισιόν πώς σκέπτεται να αντιμετωπίσει την πρόταση που έγινε από την Κομισιόν να προταχθούν οι πληρωμές για, πολλές, για πολλά διαφθορτικά ταμεία για τις πιο ευάλωτες χώρες. Αυτές που έχουν λάβει δηλαδή ενισχύσεις από τον μηχανισμό σταθεροποίησης έχει προτείνει ο Μπαρόσο και η Κομισιόν να προταχθούν πληρωμές 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2012 από όλα τα διαφθορτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, το Κοινωνικό το περιφερειακής ανάπτυξης, ακόμα και της αλίας σε κάποιο μικρό βαθμό. Πώς αντιμετωπίζουμε την πρόταση αυτή. Θα κάνουν διορθωτική επιστολή για τον προϋπολογισμό ή πάντως πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Διότι αυτά είναι επιπροσθέτως των πληρωμών που προτείνονται ήδη στο σχέδιο προϋπολογισμού. Τότε, στην περίπτωση λοιπόν αυτή, έχουμε κάποιο πρόβλημα, διότι πρόκειται για σχεδόν 3 δισεκατομμύρια σε πληρωμές παραπάνω. Είναι περίπου 2,5% αύξηση πολιτικά λοιπόν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, του συνόλου των πληρωμών. Απάντηση παρακαλώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι και αυτό πρέπει να ενταχθεί μέσα στο συνολικότερο πλαίσιο. Η Κομισιόν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση. Κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις επιπτώσεις της πρότασης που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση σε ποσοστό, αυτή είναι η πρόταση. Η πρόταση στόχο έχει να είναι κάτι σε θελούσια βάση από πλευράς κρατών μελών. Επομένως τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο και θα αποφασίσουν κατά πόσον θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα και ε, τι ποσό απαιτείται. Οι δυνατικά λοιπόν ε, μέγιστες επιπτώσεις πληρωμής θα είναι μέχρι και 6 δισεκατομμύρια για το 2012, αλλά ε, αυτό είναι το μέγιστο όριο ανάλογα με τα αιτήματα. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι αυτή η στιγμή για να ζητήσει επιπλέον πληρωμές ε, γιατί πρέπει να επιβεβαιωθούν είτε υλοποιηθούν είτε όχι. Η βασική ε, υπόθεση που είχαμε και είχαμε και στην επιστολή και τις κοινέ δηλώσεις για τις πληρωμές, ιδίω για την κατηγορία 1β, είναι ότι εάν υπάρχουν ανάγκη για επιπλέον ε, πληρωμές στη διάρκεια του έτους θα υπάρχει δυνατότητα μέσω διορθωτικού προπολογισμού να ζητηθεί αύξηση στις πληρωμές. Προς το παρόν έχουμε διαπιστώσει ότι το πνεύμα αυτής της κοινή δήλωσης δοκιμάζεται στη διάρκεια του 2011 θα δούμε πώς θα πάει η εφαρμογή και για να απαντήσουμε και στις άλλες σας ερωτήσεις, η εφαρμογή και για την έρευνα και για την πολιτική συνοχή πηγαίνει ως αναμένεται, δεν υπάρχει πρόβλημα κατά την εκτέλεση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξετάσει τα αιτήματα για πληρωμές σε όλες τις γραμμές προπολογισμού και να δει τι ε, υποχρεώσεις υπάρχουν, θα κάνει και προτάσεις για προσαρμογές και από αυτής της βάσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δει κατά πόσον ε, οι κατάλληλες υποχρεώσεις, ε, αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2011 επαρκούν. Μία σύντομη παρατήρηση ως προς την απάντηση. Σε ό,τι φορά αυτές τις κοινέ δηλώσεις. Μέχρι στιγμής δεν ήταν και πολύ επιτυχημένες. Δεν με καθησυχάζει λοιπόν ότι θα είναι χέγγιο παροχή των απαραίτητων πληρωμών. Είναι κάπως ασθενές αυτό το μέσο των δηλώσεων. Και αν πραγματικά φιλοδοξούμε να εξασφαλίσουμε 2,5 με 3 δις ε, πληρωμές και μάλιστα σε front load από πολιτική άποψη είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε περισσότερα κονδύλια στην Πορτογαλία, την Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δεν είμαι βέβαιος, δεν έχω πιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξασφαλίσει τα πολιτικά εχέγγυα και είναι σίγουρη ότι θα βρει αυτά τα επιπλέον κονδύλια. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε λύση. Αμφιβάλλω αν είναι το σωστό εργαλείο οι δηλώσει. Έχω και εγώ ένα προβληματισμό και ένα ερωτηματικό. Ναι, με να επιταχύνουμε τις πληρωμές, αλλά μόνο τα καταφέρουμε. Όχι με τους πρώτους έξι μήνες να επιταχύνουμε τις πληρωμές και μετά να σταματήσουν όλα. Και αμφιβάλλω για την ικανότητά μας να εκτελέσουμε τα σχέδια με τόσο εκλεπτισμένο τρόπο που θα μας επιτρέψει να τα αξιοποιήσουμε και να επιτύχουν. Ε, μας ενδιαφέρει φυσικά η πρόταση Μπαρόζο και υπευλήθησε πολύ κατάλληλη συγκυρία. Αν θέλουμε όμως να δοθεί συνέχεια θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια αυτή και να τη διαφυλάξουμε. Δεν αρκεί η κοινή επιστολή που είχαμε πέρυσι και που δεν απέφερε και καρπούς. Ο κύριος Γκοτμάνης ένα σύντομο σχόλιο στην, Επιτροπή, στην Περιφερειακή Επιτροπή. Μιλήσαμε με τον Επίτροπο Χάν και οι συνάδελφοι από την Ελλάδα και άλλες χώρες ρώτησαν το εξή στον Επίτροπο Χάν, που είναι αρμόδιος για τα περιφερειακά θέματα. Μήπως θα μπορούσετε ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης να μας δώσετε τα, τα χρήματα τώρα? Τότε είπε ο Επίτροπος ότι θα πρέπει να δείτε να κοιτάξετε άλλα προγράμματα γιατί δεν θα σας δώσουμε επιπλέον κονδύλια. Αν, θέλουμε, αν θέλετε προκαταβολή των χρημάτων της χρηματοδότησης, τότε θα πρέπει να είστε ε, ικανοί να αναδιαρθρώσετε όλα σας τα προγράμματα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι τέτοιες προτάσεις είναι και επικίνδυνες. Να πούμε θα προκαταβάλουμε 2-3 δισεκατομμύρια για διαφορετικές πιθανότητες. Αν παραμείνουμε στη χρηματοδότηση, τότε χρειαζόμαστε και εγγυητική επιστολή από τι αρμόδιες για το προπολογισμό αρχέ από όλα τα κράτη-μέλη, ότι αυτοί που έλαβαν τα κονδύλια θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση. Αλλιώ θα πούμε ανάληψη υποχρεώσεων ναι, πληρωμέ όχι. Και θα μα μείνουν 2-3 δισεκατομμύρια ε, σε υποχρεώσει που δεν έχουμε εκπληρώσει. Και από άποψη δημοσιονομική πειθαρχία, κάτι τέτοιο θα είναι επίση επικίνδυνο. Καλά, ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γύρο της ε, συζητήσεως. Για το ίτερ τώρα θα πω το εξής. Έχουμε συζητήσει, συζητήσαμε μάλλον και με τους συντονιστές. Εδώ πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, αφενός το πρόβλημα του ποσού που θα μπει στην συνήθη χρηματοδότηση του προγράμματος ίτερ για τον προπολογισμό 2012 και εδώ πρέπει να λάβουμε θέση σχετικά με το τι θα εγγράψουμε στον προπολογισμό 2012. Εκ παραλλήλου, εξακολουθούμε να έχουμε επιτάπητο την ε, πρόταση μεταρρύθμισης του ε, ισχύοντος πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου από, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγχρηματοδότηση του ΙΤΕΡ. Θα θυμάστε ότι ήταν και στη δέσμη διαπραγματεύσεων του ε, τέλος του περσινού έτους και όπου τελικά δεν είχαμε συμφωνήσει. Το θέμα αυτό θα επανέλθει πιθανόν το, μέσα στο φθινόπωρο διότι ο στόχος πολιτικά της Πολωνικής Προεδρίας είναι να καταλήξει σε νέα θέση του Συμβουλίου για την χρηματοδότηση αυτού του πλεονάσματος δαπανών της τάξης του 1 περίπου 3 δισεκατομμυρίου ευρώ για τα ίτερ τροποποιώντας τη δημοσιονομική προοπτική. Εμείς κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου. Για τον κίνδυνο να αναμειχθεί η συζήτηση φέτος για τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου 2012 με την μελλοντική χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ, ενώ θα πρέπει τα θέματα αυτά να παραμείνουν ξεχωριστά. Οι υπόλοιπε ομάδες πλήν των πρασίνων είναι υπέρ. Εμείς ωστόσο θέλουμε να αποφύγουμε να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών πτυχών των διαπραγματεύσεων και να αναμειχθούν σε ένα πακέτο. Το λέω λοιπόν εδώ δημοσία για να το ακούσει και η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Προς Θεού μη μας φέρετε σε μια θέση όπου την πρώτη μέρα της συνδιαλλαγής στις 8 Νοεμβρίου να έχουμε δύο θέματα, τη συμπλήρωση χρηματοδότηση του Ίτερ και τον προπολογισμό του 2012, διότι τότε θα έχουμε το πακέτο, τη σύγκρουση και δεν θα μπορέσουμε να ε, κάνουμε σωστά τη συζήτηση. Ας φτιάξουμε λοιπόν τα χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να παραμείνουν ξεχωριστά τα θέματα αυτά και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετική συμφωνία. Τέλος, θα ήθελα να αποτελέσω φερέφωνο του, της εισηγητρίας μας για να ζητήσω από όλα τα μέλη να την βοηθήσουν να κάνει τροπολογίες αρνητικής προτεραιότητας. Διότι δεν έχει τέτοιες. Υπάρχει έλλειψη τέτοιων και η συνεδρίαση που έγινε προημερών με τους εισηγητές των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό καταλήγουν οι περισσότερες και χωρίς να προτείνουν ιδιαίτερα παραπάνω δαπάνες να επανέλθουμε στις, στα νούμερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θέλουμε όμως να είμαστε σοβαροί, να μην υπερβούμε το κατόφλιο και κυρίως στις κατηγορίες 1α και 4 ή να μην το υπερβούμε υπερβολικά, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή με εύλογο τρόπο το μηχανισμό ευελιξίας και αν ταυτόχρονα θέλουμε να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες θα πρέπει να έχουμε και αρνητικές προτεραιότητες, να έχουμε το θάρρος να πούμε θέλω περισσότερα για την διαβίου κατάρτιση για την Παλαιστίνη, αλλά αφαιρώ από το ΑΒ ανάγκη την υποστήριξή σας, διότι θα είναι δύσκολη η συγκέντρια αλλά εάν θέλουμε να επιτύχουμε την απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία, θα πρέπει να αρχίσουμε να τα στοχαζόμαστε αυτά. Κυρία Συγκήτρια, θέλετε να ολοκληρώσετε. Δύο λόγια μόνο. Ευχαριστώ για όλες σας τις παρεμβάσεις. Ε, νομίζω ότι συζητήσαμε ε, πράγματα πολύ χρήσιμα και εις βάθος και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε περιμένω την απαραίτητη συνεισφορά σας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σίγουρα τις κατηγορίες 1α και 4. Ευχαριστώ πολύ. Je vous remercie. Alors je crois que nous avons épuisé l'ordre du jour. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Ούτε ή άλλο είναι και γκρέσλε δεν ε, μπορεί να έρθει, σήμερα, ε, να έρθει. οπότε το αναβάλουμε το θέμα της για άλλη φορά. Ραντεβού στο Στρασβούργο, Δευτέρα στις 7 για μια πραγματικά μακροσκελή ψηφοφορία. Δυόμιση ώρες θα κρατήσει. Φέρετε, να φέρετε μαζί σας ποτό, τις κάρτες ψηφοφορίας και την καλή σας διάθεση γιατί μας περιμένει δύο ψηφοφορία για το δημοσιονομικό κανονισμό.